ο κρατικός φόνος γυναικών και άλλων ε, ανθρώπων που θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Ήταν ο τελευταίος ομιλητής στον γύρο αυτό ομιλιών ενός λεπτού και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Θωμά Μαν για τη δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Και δίνω το λόγο στον κύριο Τόμας Μαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει δώσει ένα σημαντικό ε, μήνυμα σε σχέση με τη δημογραφική αλλαγή. Πρώτη φορά υπάρχει ένα νέο πακέτο το οποίο καλύπτει και τους νέους και τους ηλικιωμένους. Πρόκειται για την ε, δικαιοσύνη μεταξύ των γενναιών. Μια νέα προσέγγιση. Ε, μιλούμε λοιπόν μαζί και όχι ο ένας εναντί του άλλου. τα μελη με, τα, με τους ισολογισμούς μεταξύ των γενεών μπορούν να έχουν μια σωστή πρόβλεψη για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθούν οι πληρωμές συντάξεων και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλειας. Με τον έλεγχο των γενναίων δημιουργείται και ένας νέος τρόπος ο οποίος μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά τα προβλήματα που έχουμε χωρίς παρενέργειες που θα επιβαρύνουν παραπάνω τις γενές. Επίσης, σε ό,τι αφορά το θέμα των συντάξεων, θα πρέπει να υπάρξει ένα, ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ενιαία ηλικία συντοξιδότησης και επίσης θα πρέπει να διατηρηθούν τα εθνικά κριτήρια για την ηλικία συνταξιδότησης. Δεν πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να υποχρεώνουν τους ανθρώπους με ένα αυθαίρετο τρόπο να εγκαταλείπουν το χώρο εργασίας. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του του Οκτωβρίου θεώρησε ότι, είναι, ότι δεν μπορεί να επιβληθεί μια υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης. Θα πρέπει οι άνθρωποι να μην θίγονται επί τη βάση της ηλικία τους. Για τους πιο ηλικιωμένους θέλουμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τα άτομα άνω των 50 ετών για να υπάρχουν τρεις στόχοι. Καταρχήν, το ποσοστό εργαζομένων των άνω των 50 θα πρέπει να ξεπεράσει το 55%. Δεύτερον, η πρόορη συνταξιοδότηση θα πρέπει να μειωθεί και να καταργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τρίτον, τα κρατημέλη θα πρέπει να δώσουν περισσότερα οικονομικά μέσα για τους ανθρώπους άνω των 60 ώστε να παραμείνουν περισσότερο στο χώρο εργασία. Επίση, στο άλλο άκρο του φάσματο για του νέου, Θέλουμε να υπάρξει μια εγγύηση για του νέου. Ο κάθε νέο, μετά από μια περίοδο ανεργία το μέγιστο τεσσάρων μηνών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει μια θέση ή άλλε δυνατότητε κατάτηση. Εδώ υπάρχει ή μια θέση μαθητείας ή αλλε δυνατοτητε κατάρτιση. Εδώ υπάρχει η, <clears throat> η αρχή να βοηθούμε αλλά συγχρόνως να απαιτούμε. Αλλά αυτό δεν είναι μονάχα ένας μονόδρομος. Θα πρέπει οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και προσόντα για να αποκτήσουν μια θέση εργασίας. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες ε, ε, εβδομάδες δέχτηκε μια πρόταση μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κήρυξε το έτος 2012 ως έτος της ενεργούς γύρανσης. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και επίσης θα πρέπει η Κομισιόν να θέσει και νέες προτάσεις κατά των διακρίσεων ώστε να υπάρξουν νέα κριτήρια για τους ηλικιωμένου και να μην αποκλείονται από τις ασφάλειες να έχουν τη δυνατότητα να νοικιάζουν αυτοκίνητα και να κλείνουν διακοπές, να μην έχουν να αντιμετωπίσουν μια γραφειοκρατία λοιπόν η οποία δεν επιτρέπει στα άτομα αυτά να λειτουργούν χωρίς αποκλεισμό από την κοινωνία. Γι' αυτό το ΕΛΚ έχει υποβάλει και μία νέα ε, πρόταση προ την κατεύθυνση αυτή. Κατά τα άλλα έχουμε συμφωνήσει στην Επιτροπή Απασχόληση μετά από μία σειρά από τροπολογίε που οδήγησαν σε 22 συμβασικέ τροπολογίε που επέτρεψαν μία συνένεση. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλου του συναδέλφου από όλα τα κόμματα για την ε, επικοδομητική του συνεργασία. Νέοι και ηλικιωμένοι μπορούμε να κινούμεθα και να εργαζόμαστε από κοινού. Ελπίζω ότι με αυτήν την ε, έκθεση για την ισότητα μεταξύ, για την μάλλον αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενναίων, μπορούμε να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαν. Έχω πολλούς ομιλητές τώρα. Στη διαδικασία Catch the Eye θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κέλλη. Συγχαίρω τον κύριο Μαν για τη σημαντικότατη εργασία του. Νομίζω ότι για τους ηλικιωμένους το σημαντικότερο είναι να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας προς την συνταξιοδότηση και προς την εργασία. Πρέπει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες για εθελοντικά σχέδια συνταξιοδότησης, προαιρετικής συνταξιοδότησης με περισσότερες επιλογές. Γνώριζα, είχα έναν συγγενή ο οποίος ήθελε να φύγει στη σύνταξη στα 65 αλλά είχε πει ότι το κάνει με ελεύθερη του επιλογή. Την ίδια επιλογή πρέπει να έχουν και όσοι θέλουν να φύγουν στα 67 κτλ. Η νεολαία στην Ιρλανδία είναι η ηλικιακή ομάδα με τη, που πλήττεται περισσότερο από την τραπεζική κρίση και η μόνη τους επιλογή είναι με ποιο εισιτήριο να φύγουν από τη χώρα γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας εκεί. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και η εργασία και η συνταξιοδότηση και όπως είπε και ο κύριος Μαν πρέπει να δοθούν τουλάχιστον μερικές περισσότερες επιλογές στους νέους. Ευχαριστούμε. Κύριε Κέλλη, κυρία Μπρίβιν Τσούτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που μας εξέθεσε από τις συστάσεις του στην εκθεσή του την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αλλά όταν μιλάμε για τους ηλικιωμένου, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε την δυνατότητα πρώιμης συνταξιοδότησης μερικοί την αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δείχνουν ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός τρόπος για να μην απολεστούν περαιτέρω θέσεις εργασίας. Διαφέρουν βέβαια τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μεταξύ των χωρών, αλλά δεν πρέπει να δοθεί ενιαία λύση για όλα. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Θωμά Μάν. Πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι τυχαίνουν πολύ κακής μεταχείρισης από τα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη. Με πολλούς τρόπους μάλιστα, όπως η ηλικιακή άνηση μεταχείρισης στους τόπους εργασίας. Και γι' αυτό στην έκθεση αυτή ζητιέται με επιμονή η σωστή εφαρμογή της οδηγίας του 2000 για την εργασία. Ευτυχώς η τροπολογία μου για την ηλικία της συνταξιοδότης έγινε δεκτή από τον εισηγητή και στην Επιτροπή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει βέβαια, αν θέλει ένα ηλικιωμένο να εργαστεί και πέραν από την επίσημη ηλικία συνταξιοδότηση, να μπορεί να το κάνει. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε το Συμβούλιο ως προς την οδηγία για την πρόσβαση αγαθά και υπηρεσίες να εφαρμόσει τις διατάξεις κατά της άνηση μεταχείρισης με βάση την ηλικία. Και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα και για την αρχική έκθεση του εισηγητή, όχι μόνο για τις δικές μου τροπολογίες. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Μαν για την έκθεσή του. Η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Δεν πρέπει μια γενιά να ζει σε βάρος των άλλων. Και είναι απαραίτητο αυτό το οποίο γίνεται σε μια οικογένεια να αντανακλάται και στα πλαίσια μιας κοινωνίας. Ε, υπάρχει κάποια ε, αλληλεγγύη η οποία θα πρέπει να ασκείται μεταξύ των γενναίων. Εμείς έχουμε κατά κάποιο τρόπο δανειστεί τα, τους πόρους που θα πρέπει στη συνέχεια να κάνουν να ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η έκθεση του κύριου Τόμας Μάν είναι για μένα μια πολύ καλή ε, έκθεση προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέιντου έχει το λόγο. Δεν θέλετε το λόγο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η κυρία Σαχνάλοβα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαγενειακή αλληλεγγύη περιγράφεται ορθότατα από τον εισηγητή μας, τον κύριο Μαν. Μία αξιοπρεπής συνταξιοδότηση είναι κάτι που πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για όλους πάντοτε. Ε, εξού και το πρόβλημα της παραγράφου 90, διότι εκεί ε, προτείνεται η αντικατάσταση ε, του αναδιανεμητικού συστήματος με ένα χρηματοδοτούμενο σύστημα συνταξιοδότησης. Έχουμε πρόβλημα με τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία που επλήγησαν τα τελευταία χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις ε, απόλυσαν πάνω από 20% της αξίας ε, των ε, στοιχείων ενεργητικού τους. Έπρεπε λοιπόν να απολύσουν με απώλειες για να επιβιώσουν αυτά τα ταμεία. Ε, με τέτοια χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, στα οποία επενδύουν αυτά τα ταμεία, πώ περιμένουμε από του πολίτε να ε, του έχουν εμπιστοσύνη για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή του ε, συνταξιοδότηση. Ο κύριος Μίκολας πάλι από τη Σλοβακία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η δημογραφική αλλαγή επηρεάζει την πυραμίδα των ηλικιών. Και λόγω αυτής της αλλαγής και του γεγονότος ότι έχουμε περίπου 1,5 παιδί για κάθε γυναίκα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό της χαμηλής γεννητικότητας. Υπάρχουν πολλά, πολλά προβλήματα στην κοινωνία που εμποδίζουν τις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε φορολογικές ελαφρύνσεις στις οικογένειες με πολλά παιδιά. Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ενεργό γύρανση. Αυτό σημαίνει να εξαλείψουμε διάκριση επί τη βάση ηλικία και στην πράξη. Θέλω να χαιρετήσω τις πολιτικές για ενεργό γύρανση που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν στη ζωή των κοινοτήτων τους και να ζουν σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης μεταξύ των γενναίων. Και τώρα θα ακούσουμε δύο Ρουμάνους ομιλητές, ξεκινώντας με την κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει μεγάλη επικαιρότητα με τους νέους και τους ηλικιωμένους που έχουν και οι δύο ομάδες του πληθυσμού πολλά προβλήματα να βρουν θέσεις εργασίας. Η ισορροπία μεταξύ των γενεών θα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στα επερχόμενα έτη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έννοια τη ασφάλειας μέσα και στην πολιτική της Ευρώπης 2020 για να μπορέσει να υπάρξει ένα επίπεδο απασχόλησης 75%. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Θεωρώ ότι τόσο η Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτήν την συμφωνία μεταξύ των δύο γενεών, των γενεών μάλλον, σαν βασικό στοιχείο, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μια αηφόρο ανάπτυξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Τέλο, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαν, γιατί κατάφερε να καθορίσει στην έκθεσή του μια σειρά από πάρα πολύ ελκυστικέ λύσει, όπω παραδείγματο το πακέτο για την ευρωπαϊκή εγγύηση απασχόληση ή κατάρτιση mm-hmm. για του νέου και το πακέτο 50 ετών και παραπάνω. Ο κ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, τα επόμενα χρόνια θα βρεθούμε αντιμέτωποι όχι μόνο με τα προβλήματα της κρίσης αλλά και με άλλες προκλήσεις, ε, κυρίως με τη δημογραφική πρόκληση και την απερίμωση κάποιων περιοχών. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κύριο ρόλο να διαδραματίσει, να εξασφαλίσει τους όρους υπό τους οποίους οι πολίτες θα δεχτούν τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις αυτών των προκλήσεων. Χρειαζόμαστε τα σωστά ε, χρηματοδοτικά μέσα, όπως παραδείγματος χάρη τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι καλό θα ήταν να εμπλακούν στα κοινά. Να επενδύσουμε λοιπόν στη νεολαία, να προσφέρουμε πρόσβαση στους νέους σε μια καλή εκπαίδευση και να δώσουμε την ευκαιρία να βρουν μια καλή θέση απασχόληση, να τους ενθαρρύνουμε να ανοίξουν ε, δικές τους επιχειρήσεις ε, έτσι θα καταπολεμήσουμε και ένα από τους παράγοντες υπογεννητικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επίτροπος Μάλμστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή, τον κύριο Μάν. Είναι πάρα πολύ καλή και διεξοδικότατη η έκθεσή του γιατί παρουσιάζει όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, σε αυτό το τομέα της δημογραφίας. Ε, έχουμε στρατηγικές τόσο ώστε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστούν για τη γύρανση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τις επιπτώσεις της. Ε, υπάρχουν, πάρα πολλές δράσεις, η εγγύηση για την νεολαία, το πρόγραμμα 50 συν, η πρωτοβουλία για την διαχείριση της γύρανσης κτλ. κτλ. Επίσης υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις ε, για να προσδιορίσουμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη την αρχή της διαγενειακής αλληλεγγύης, γιατί είπατε και εσείς σωστά ότι είναι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, η Επιτροπή έχει εγκρίνει δύο βασικές πρωτοβουλίες. Ήδη έχουμε την πράσινη βίπλο για τις συντάξεις και του χρόνου θα ακολουθήσει η λευκή βίπλος για τις μελλοντικέ δραστηριότητες τη Ένωσης και επί τη βάση της πρότασής θα ορίσουμε το 2020 ως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γύρανση. Επίσης θα υποβάλουμε την έκθεσή μας για την δημογραφική ε, πρόκληση και θα δούμε πώς ε, έχουν πληγεί τα κράτη-μέλη από την ε, κρίση και κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Γιατί τις επόμενες δεκαετίες μην ξεχνάτε ότι θα φτάσουν στη σύνταξη τα παιδιά του baby boom και μην ξεχνάτε ότι οι νέες γενιές Ευρωπαίων θα προέρχονται παραδείγματος χάρη ίσως από τρίτες χώρες και έτσι θα χρειαστούν ε, νέες πολιτικές ε, στα κράτη-μέλη. Ε, μόνο για να επιτύχουμε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της δημογραφικής γύρανσης μέσω της ενεργούς γύρανσης με της βελτίωσης κατάστασης των νέων μέσα στην αγορά εργασίας, της ένταξης των μεταναστών, να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα για λόγους εργασίας και σε όλα σε όλο αυτό το πελώριο έργο προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία φυσικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε. Ε, συνάδελφοι, λίγη η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Και τώρα περνούμε στην τελευταία έκθεση της ε, σημερινής.